Κύριε και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, σα καλησπερίζω στην ιδρυτική μα συνεδρίαση τη Υποεπιτροπή Ασφαλεία και Άμυνα. Συγχαίρω όλους που εξελέγησαν και επανεξελέγησαν. Η Υποεπιτροπή μας δεν εννοεί ότι είναι δεύτερης κατηγορίας επιτροπή αλλά μια επιτροπή συζήτησης όχι για θέματα που δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά όπως η άμυνα αλλά για στοχεύει σε, μια επιτρο... σε δημιουργία μιας κοινή πολιτικής άμυνας που προβλέπεται από τις συνθήκες. Και η προηγούμενη θητεία μας έδειξε ότι προσπαθούμε να τα υλοποιήσουμε όλα αυτά. Ελπίζω το ίδιο να γίνει και σε αυτή τη θητεία. Αρχίζει λοιπόν αυτή η συνεδρίαση. Σήμερα θα εκλέξουμε το προεδρείο μας, δηλαδή τον πρόεδρο και τις, τους αντιπροέδρους. Για να δούμε λοιπόν για τον πρόεδρο. Α, να σας πω και ποιοι είναι οι αναπληρωματικοί που έχουν σήμερα δικαίωμα να ψηφίσουν γιατί αντικαθιστούν πλήρη μέλη. Για τους σοσιαλιστές έχω τον κύριο Βικτόρ Μποστινάρου που θα αντικαταστήσει, που θα ψηφίσει και για το ΕΛΚ τον κύριο Ιβο Μπελέτ, τους κυρίους Ιβο Μπελέτ και Μακάλιστερ. Η απαρτία είναι 8 βουλευτές. Υπάρχει λοιπόν απαρτία. Αρχίζουμε λοιπόν με τις υποψηφιότητες. Ποιες πολιτικές ομάδες θέλουν να προτείνουν υποψηφιότητες. Ο Τζέφρι Βανόρντεν. Όρντεν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Χαρήκαμε πολύ την προηγούμενη Προεδρία σας της Υποεπιτροπής. Εξ των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών προτείνω την κυρία Άννα Φωτσίγκα ως πρόεδρο της υποεπιτροπής. Η κυρία Φωτσίγκα είναι πολύ εξέχον μέλος του Πολων, της Πολωνικής Βουλής. Ήταν επικεφαλής της ε, Πολωνικής Προεδρίας του πρωτοκόλου της Πολωνίας και έχει επομένως τεράστια εμπειρία για τη θέση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κυρία Φωτίγκα, δέχεστε την υποψηφιότητά σας. Ναι, τη δέχομαι. Ευχαριστούμε. Η κυρία Φωτσίγκα είναι πλήρες μέλος της Υποεπιτροπής και έχει συμπληρώσει τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων, πληρεί λοιπόν τα προσόντα. Υπάρχει καμία άλλη υποψηφιότης. Άννα Γκόμες. Ναι, Πρόεδρε, και εγώ σας ευχαριστώ για την εξαιρετική προεδρία της Υποεπιτροπής στην προηγούμενη θητεία. Θέλω να υποβάλω ατομικά την υποψηφιότητά μου, προσωπικά μάλλον. Δεν αμφισβητώ την ποιότητα της υποψήφιας που ανέφερε ο κύριος Βαν Όρντεν, της κυρίας Φωτίγκα, αλλά νομίζω ότι η ομάδα του πάντοτε προάσπιζε θέσεις που αμφισβητούσαν την αναγκαιότητα μιας πολιτικής κοινή άμυνας και ασφαλείας. Αν αυτή λοιπόν είναι η γραμμή της επόμενης Προεδρίας, τότε νομίζω ότι αυτό δεν αρμόζει καθόλου στην υποεπιτροπή μας. Εγώ είμαι μέλος της υποεπιτροπής αυτής από τη δημιουργία της το 2004 Γνωρίζω πολύ καλά πόσα έχουν γίνει από τα μέλη της για να αυξηθεί η αξιοπιστία της, καταρχήν υπό την προεδρία του κυρίου Φων Φόγκαου και μετά από εσά. Και πιστεύω ότι, ίσως να μας το εξηγήσει η κυρία Φωτεγκάλα, εάν η κυρία Φωτέγκα συμμερίζεται τις ίδιες θέσεις με τον συνάδελφό της κύριο Βανόρντεν που την πρότεινε, και που ανέκαθεν και με μεγάλη συνέπεια προάσπιζε τη θέση κατά της δημιουργίας μιας Ευρώπης ασφαλείας και άμυνας, τότε νομίζω ότι δεν θα ήταν αρμόζον να βάλουμε στην Προεδρία τέτοιες θέσεις, ανθρώπους που αντιπροσωπεύουν τέτοιες θέσεις, ιδίως σε αυτή την περίοδο κρίσης που θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο η άμυνα και η ασφάλεια. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την κυρία Φωτίγκα αν μπορεί να μας εξηγήσει αυτό το πρόβλημα. Αν συμμερίζεται δηλαδή τις ίδιες θέσεις με τον κύριο Βανόρντεν που την πρότεινε. Τότε, σε αυτή την περίπτωση, θέλω και εγώ να είμαι υποψήφια και με μυστική ψηφοφορία. Δύο σημεία πρώτον για την πιθανή παρουσίαση υποψηφιωτήτων. Υπάρχει η δυνατότητα αυτή. Πρέπει η υποψηφιότητα να γίνει είτε εξ ονόματος ομάδας, είτε να προταθεί υποψηφιότητα από δύο βουλευτές, γιατί απαιτείται το 5% των μελών. Αν υποστηριχθείτε στην πρωτοβουλία σας από δύο βουλευτές, έχετε το δικαίωμα να είστε υποψηφία. Αυτά επί της διαδικασίας. Σε, πολιτικό επίπεδο θα δώσω το λόγο στην ομάδα των συντηρητικών η οποία κατέθεσε την υποψηφιότητα, η κυρία Φορτιγκά Ή μάλλον ο κύριος Βανόντεν. Δεν είναι δική μου υποψηφιότητα. Είναι, είναι μια πρόταση της πολιτικής μου ομάδας Δεύτερον, βρισκόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι ένα δημοκρατικό κοινοβούλιο, εκπροσωπεί έθνη και πολιτικές απόψεις διαφορετικές και θα πρέπει οι απόψεις αυτές να εκπροσωπούνται όλες. Και τρίτον, οι προτάσεις ορισμών, διορισμών βασίζονται στο σύστημα αντεχόντ, το οποίο ε, θα έλεγα διασώζει τα συμφέροντα των μικρών ε, πολιτικών ομάδων και των μικρών χωρών ακόμα και θα ήταν πραγματικά πολύ επικίνδυνο να ακολουθήσουμε μια διαφορετική κατεύθυνση, αλλά νομίζω ότι η κυρία Φορτίγκα η Ιδία θέλει το λόγο. Uh, I do represent... Uh, Πράγματι εκπροσωπώ την Πολωνία. Την εκλογική, είναι η εκλογική μου περιφέρεια. και ήμουνα υπεύθυνη για την πολωνική αντιπροσωπεία στη διακυβερνητική διάσκεψη κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης της συνθήκης της Λισαβόνας. Και γνωρίζω καλά το άρθρο 42, το οποίο ασχολείται με τα θέματα της ΚΕΠΑ και γι' αυτό θα ήθελα να εκφράσω την άποψή μου και το γράμμα και το πνεύμα της συγκεκριμένης αυτής νομικής ρύθμισης ορίζει την ΚΕΠΑ και ιδιαίτερα το άρθρο 2 χωρίς καμία διάκριση εις βάρος κρατών μελών, τα οποία επιζητούν και αυτά την δική τους ασφάλεια με διαφορετικές συμμαχίες όπως το ΝΑΤΟ. Και μιας και εγώ ήμουν μέλος και της αντικομουνιστικής επανάστασης αντιπολίτευσης στην Πολωνία εμείς εκτιμούμε ιδιαίτερα και εγώ η Ιδία εκτιμώ ιδιαίτερα την ασφάλεια που μας παρέχει το ΝΑΤΟ. Μετά από διαπραγμάτευση επικυρώθηκαν οι ρυθμίσεις αυτές από την Πολωνική Βουλή, υπεγράφει από τον Πολωνό Πρόοδο και αυτό με υποχρεώνει νομικά να το στηρίξω. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση η ΚΕΠΑ στην περιοχή την οποία εγώ εκπροσωπώ να αντικαταστήσει την προστασία που παρέχει το ΝΑΤΟ. Καλώς, σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Ο κύριος Πάσκου μια τελευταία λέξη διαδικαστικά Εγώ θα υποστηρίξω την υποψηφιότητα της κυρίας Γκόμες, οι άλλοι θα πούνε τις απόψεις τους, αλλά η ουσία ποια είναι. Δεν είναι οι προσωπικές, ε, αν θέλετε, απόψεις των υποψηφίων. Είναι οι στάσεις ε, την οποία κρατούν σε μια επιτροπή που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν εμείς περιφρονήσουμε αυτή την πολιτική στην Επιτροπή η οποία η, την δημιουργεί κατεξοχήν, την στηρίζει και την προωθεί κατεξοχήν. Και αν τα μεταφέρουμε όλα στο ΝΑΤΟ, κάτι το οποίο υποστηρίζω, εγώ ήμουνα υπουργό Άμυνα και διαπραγματεύτηκα την ένταξη της Ρουμανίας στο ΝΑΤΟ. Είμαι υπέρ του ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα όμως δεν δέχομαι εγώ ότι είναι ή το ένα ή το άλλο, ότι είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Θεωρώ ότι συμπληρώνουν το ένα το άλλο. Κοιτάξτε, αν κατάλαβα κάτι τέτοιο από αυτά που είπατε δεν θα είχα ζητήσει το λόγο, αλλά δεν το κατάλαβα. Κοιτάξτε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτές τις θα τις κάνουμε. Πέντε χρόνια στην Επιτροπή μας. Έτσι δεν είναι, Τζέφρι, αγαπητέ Τζέφρι. Προτείνω λοιπόν να περάσουμε στην ε, διαδικασία μας και να ψηφίσουμε είτε διαβοής, ε, εάν είναι μόνη υποψήφια η κυρία Φωτίγκα, είτε με ψηφοδέλτιο ή μυστική ψηφοφορία ηλεκτρονική, εφόσον η κυρία Γκόμες εμένει στην ε, υποψηφιότητά της. Μάλιστα, αν επιμένεις, ωραία, μυστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, παρακαλώ να λάβετε όλοι σας τις κάρτες για να ψηφίσετε. Η κυρία Γκόμες έχει καταθέσει υποψηφιότητα. Την υποστηρίζουν πάνω από δύο μέλη της Υποεπιτροπής. Άρα είναι νόμιμη, νομότυπη υποβολή της υποψηφιότητας. Είναι μέλος της Επιτροπής μας. Έχει καταθέσει σχετική δήλωση ε, οικονομικών συμφερόντων, Άρα είναι αποδεκτή, παραδεκτή η αίτηση, η υποψηφιότητα και παρακαλώ ψηφίζουμε με μυστική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έχουμε τα δύο, τα δύο κουμπιά, το συν και το πλήν. Το πράσινο κουμπί για λόγους αλφαβητικής σειράς. Το πράσινο θα αντιστοιχεί στην κυρία Φωτίγκα. Αν ψηφίσετε την κυρία Φωτίγκα θα πρέπει να πατήσει το πράσινο κουμπί ενώ αν ψηφίσετε με το μείον, το κόκκινο δηλαδή κουμπί, θα ψηφίσετε για την κυρία Γκόμες. Ήταν κατανοητό αυτό για τους πάντες. Άρχεται η ψηφοφορία. Έχουμε δύο υπεράριθμους. Ας ψηφίσουν πρώτα τα τακτικά μέλη και να υπολογίσετε αν χρειάζονται να πληρωματικά. Έχουμε δύο υπεράριθμους. Il me reste ακόμη υπεράριθμό. Δεν μπορώ να σα πω από ποια ομάδα. Το καλύψατε. Υπενθυμίζω την σύνθεση των ομάδων για να μπορέσει ο καθένας να κάνει τον υπολογισμό του. Εννέα ψήφους έχει το ΕΛΚ. Σοσιαλιστές Δημοκράτες 8 συντηρητικοί μεταρρυθμιστέ 3, φιλελεύθεροι 3, η Γκουε 2, η Πράσινη 2, η Ευρώπη των Ελευθεριών και των Δημοκρατιών 1 και μείνει γεγραμμένη μία ψήφο και παραμένει μία υπεράριθμη ψήφος. Αν θέλετε βγάλτε τις κάρτες σας. Εκείνοι που δεν ψηφίζουν να βγάλουν τις κάρτες του από το μηχάνημα. Πρέπει να βγάλετε την κάρτα από το μηχάνημα. Τώρα είμαστε εντάξει. Όχι, 32. Λοιπόν, για κάθε πολιτική ομάδα να γίνει η επαλήθευση, παρακαλώ, γρήγορα. Τώρα είμαστε 30. Είναι σωστά τα νούμερα. Αρχή η συνεδρίαση λοιπόν με 30 βουλευτές. Ψηφίσαν όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Όχι, ξαναγυρνάμε στους 31. Ε, δεν νομίζω να είναι περίπλοκο αυτό που σας λέω. Καλά που δεν είμαστε και 250. Ξανά αρχίζει η συνεδρίαση. Πράσινο η κυρία Φωτίγκα, κόκκινο η κυρία Γκόμες και παραμένουν οι 31 κάρτες στα μηχανήματα. E, Το έλκει είναι εντάξει μαζί με μένα, με υπολογίσατε μένα. Οχτώ ψήφισε οι σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ωραία. Λοιπόν, έχω 30 ψηφίζοντες τώρα. Κυρίσω το πέρας της ψηφοφορίας και το αποτέλεσμα είναι 15 υπέρ της κυρίας Φωτίγκα και 8 υπέρ της κυρίας Γκόμες. La majorité était à 15, donc Madame Fotiga est élue. Με την πλειοψηφία λοιπόν 15 ψήφων η κυρία Φωτίνκα εκλέγεται και της παραδίδω την Προεδρία. Mm-hmm. I would like to, thank Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Υποεπιτροπή. Υποεπίτροπη. Ασφάλειας και άμυνας που με εξέλεξε σε αυτή την θέση της Πρόεδρου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον απερχόμενο πρόεδρο για την εξαιρετική δουλειά του και ασφαλώς υπόσχομαι ότι θα στηριχθώ και στη δική του εμπειρία αλλά και στην εμπειρία της γραμματείας. Και τώρα θα περάσω στο σημείο 2 της ημερήσιας διάταξης για σήμερα. Θα θέλαμε να ψηφίσουμε λοιπόν τώρα αντιπροέδρους της Υποεπιτροπής. Απαρτία υπάρχει. Ισχύουν οι ίδιες αντικαταστάσεις των τακτικών μελών από αναπληρωτές. Και καλό τους εκπροσώπους των ομάδων να προτείνουν υποψηφίους για τη θέση πρώτου Αντιπρόεδρου της Υποεπιτροπής. Κύριε Κέλλαμ, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια σας. Εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της ομάδας του Ευρωπαϊκού Ευρωπαϊκό δεν θέλω να υποβάλω τον Μιχαήλ Γκόνερ ως υποψήφιο για τη θέση του πρώτου αντιπροέδρου. Έχει εντυπωσιακή εμπειρία από την ε, πολιτική εξωτερικής εξωτερικών υποθέσεων και άμυνας και έχει κάνει πολύ καλό έργο. Έχει επιδείξει μεγάλη διάθεση για συνεργασία και συμβασμούς. Προτείνουμε λοιπόν τον κύριο Γκόνερ. Είναι αποδεκτή η υποψηφιότητα κύριε Γκόνερ. Γκάιερ. Καλώς έχετε καταθέσει το, τη δήλωση οικονομικών ε, συμφερόντων. Σας υποστηρίζει η ομάδα σας. Προτείνω λοιπόν να εκλεγεί ο πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής διαβοής. Thank you. And therefore uh, Vice Chair. Please uh, join us. Εξελέγετε λοιπόν και περάστε παρακαλώ στο Προεδρείο. Δεύτερο αντιπρόεδρο έχει επίσης προτείνει μία ομάδα. Παρακαλώ. Για τον κύριο Τιτσινό. Κύριε Κέλλεμ, Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της ομάδας μου θα ήθελα για τη θέση του δεύτερου αντιπροέδρου της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας να προτείνω τον κύριο Γιάννου Στέντιγκερ που κάθεται εκεί πίσω. Κύριε Σέτινα, δέχεστε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 as second vice chair of subcommittee and please join us here at the table. Now, please. Και τώρα παρακαλώ. Εκ μέρους των Σοσιαλιστών Δημοκρατών, να μας προτείνετε υποψήφιο για τη θέση του τρίτου αντιπροέδρου της Υποεπιτροπής. Κυρία Πρόεδρε, ο κύριος Παστσού. Θα ήθελα να υποβάλω την υποψηφιότητα κυρίου Κάτσου ως υποψηφίου για τη θέση του τρίτου αντιπροέδρου. Έχει μεγάλη ε, εξειδικεύση και εμπειρία στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Η δήλωση οικονομικών σφαίρων έχει κατευθεί. Ο κύριος Καν δέχεται την υποψηφιότητα. Έκτος μικροφώνου. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ να επικυρωθεί η υποψηφιότητα αυτή. Δια δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος. Σας ευχαριστώ. Και τώρα η τελευταία και τέταρτη υποψηφιότητα για τη θέση τέταρτου αντιπροέδρου εκ μέρου τη ε, πολιτική ομάδα τη ΓΚΟΕ. Παρακαλώ, εκ μέρου τη ΓΚΟΕ, ποιο θα λάβει το λόγο για να προτείνει υποψήφιο. Από την ΚΟΕ θα θέλαμε να προτείνουμε την κυρία Λόζινγκ. Είναι από το 2009 βουλευτής, ήταν συντονίστρια της ομάδας κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περίοδου. Ήταν επίσης και ε, συντονίστρια της ομάδας μας και αυτό δείχνει ότι είναι εμπειρογνώμων γενικά στα θέματα της ασφάλειας και της άμυνας και την προτείνουμε για την τέταρτη αντιπροεδρία. Λοιπόν, δέχεστε την υποψηφιότητα. Η δήλωση των οικονομικών συμφερόντων έχει κατατεθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως εκ τούτου. Μπορούμε να εκλέξουμε λοιπόν την Αντιπρόεδρο διαβοής. Thank you and please join uh, Μπορείτε να έλθετε και εσείς στο Προεδρείο. Thank you. Now we Καλώς. Περνάμε στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης. Θα ήθελα να επιβεβαιώσουμε το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεών μας. Μέχρι το τέλος του 2014. Η πρώτη συνεδρίαση θα γίνει στις 11 Σεπτεμβρίου. already, um, uh, already after vacations and have certainly Έχουμε πολλά θέματα μετά από τις διακοπές. Θα έχουμε πολλά θέματα μετά τις διακοπές. Εν τω μεταξύ θα μπορέσουμε να προετοιμαστούμε επίσης καλύτερα Έχουμε και το θέμα της προετοιμασίας της επόμενης συνάντησης κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουαλία. Και θα ήθελα να ζητήσω από τα μέλη του Διευρυμένου Προεδρείου να συναντηθούν στο Στρασβούργο έτσι ώστε να συζητήσουμε κάποια σημαντικά θέματα για τις εργασίες της Επιτροπής μας. Εφόσον συμφωνείτε λοιπόν με την πρότασή μου και δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσεις, δεχόμαστε την ρύθμιση αυτή σχετικά με τη συνεδριάση μας. Αυτά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο και κυρίσω το τέλος της συνεδρίασης. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την εκλογή των μελών του Προεδρείου μας.